Il Presidente. Eccoci qua. Come andiamo? La seduta è aperta. Άρχεται η συνεδρίαση. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Το πρώτο σημείο στη μερίσια διάταξη προβλέπει την παρουσίαση του προγράμματος των δραστηριοτήτων της Κροατικής Προεδρίας, δηλώσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το συμβατικό τρόπο εγγραφής είτε τον ηλεκτρικό τρόπο εγγραφής για να συμμετέχετε στη διαδικασία Catch the Eye και για να υποβάλλετε ερώτημα μέσω της μπλε κάρτας. Δίνω ευθύ λοιπόν αμέσω το λόγο στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου Πλένκοβιτσα ε, για να μας κάνει την παρουσίασή του. Σα ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Ντάβιτ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδροι, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, αξιότιμη Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμοι συνάδελφοι, νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση που βρίσκομαι εδώ σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της πρώτης Κροατικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Κροατία και τους συμπολίτε μου πρόκειται για μια ιστορική στιγμή. Μόλις πριν από 30 χρόνια έγιναν στην Κροατία οι πρώτες ελεύθερες εκλογές. Και έτσι, μετά από 9 αιώνες, ο κροατικός λαός ανέκτησε και πάλι την κυριαρχία του και η Κροατία επέστρεψε στον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη. Και χαίρομαι ιδιαίτερος που σήμερα, παραμονές της 28ης επαιτίου της Διεθνούς Αναγνώρισης της Κροατίας, τότε που τα κράτη-μέλη, τωρινά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισαν την Κροατία, εγώ έχω την ευκαιρία να εκφωνήσω ομιλία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα την αναγνώριση την επιτύχαμε σε δύσκολε περιστάσει μια επίθεση ε, πολεμική. Και χάρη στου αγωνιστέ μα, ε, η Κροατία αμήνθηκε, πριν από 25 χρόνια απελευθερώθηκε, κατόπιν ανανεώθηκε και κινήθηκε στο δρόμο τη ανάπτυξη, του εκδημοκρατισμού και τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και πριν από 6,5 χρόνια, κατέστηκε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και μάλιστα για πρώτη φορά κρατάει το πιδάλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την πορεία η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ήταν για την Κροατία στεναρός και ξεκάθαρος οδηγός σε όλες τις προσπάθειες και όλες τις μεταρρυθμίσεις που υλοποίησαμε. Χαίρομαι για την επιτυχή συνεργασία που θα έχουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το επόμενο εξάμεινο, γιατί αυτό επιθυμούν οι πολίτες μας να δείξουμε ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν απτά ωφέλη. Έχουμε λοιπόν ενώπιόν μας πολύ σημαντικές αποστολές και καθήκοντα. Καταρχήν, κυρίε και κύριοι, μία συμφωνία για το νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Μία έγκαιρη συμφωνία για το σύνολο του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου για τα επόμενα 7 χρόνια είναι προτεραιότητά μα. Και γι' αυτό το ΠΔΠ θα πρέπει να ανταποκρίνεται στι προσδοκίε όλων των πολιτών σε όλα τα κράτη-μέλη μα. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις πολιτικές συνοχής και γεωργίας, αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει τις πολυάριθμες νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συνοχή και την ενότητά μας, με σεβασμό όμως όλων των διαφορών μας, των οικονομικών, κοινωνικών και δημογραφικών. Ταυτόχρονα θα πρέπει να καταστήσει την Ευρώπη πιο αποτελεσματική και ορατή στο παγκόσμιο προσκήνιο. Και για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να δράσουμε πάρα αυτά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021. Οι μη θα απογοητεύσουμε τους πολίτες μας. Μαζί λοιπόν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συνεχίζει τις διαβουλεύσεις για το ΠΔΠ στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, δεν θα αφιστούμε προσπαθειών για να επιτύχουμε την ολοκλήρωσή της κατά την, προετοιμασία, κατά την Προεδρία μας. Έτσι θα ολοκληρώσουμε το σύνολο του νομοθετικού πακέτου για το ΠΔΕΛΤΑΠΗ και σε αυτό προσβλέπουμε σε στενή και αποτελεσματική συνεργασία με όλες τις επιτροπές και τους εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή μας την προσπάθεια. Αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε όλες τις ανησυχίες σας, τα μηνύματα και τις προσδοκίες σας. Βέβαια, κατά τη γνώμη μας, είναι κέρια σημασίας να συνεχίσουμε τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να προωθούμε ταυτόχρονα όλα τα επιμέρους θέματα. Και σε αυτό μας ενώνει ο κοινό μας στόχος, γιατί η αποτυχία μας θα ενισχύσει εκείνους που δεν επιθυμούν μια ισχυρή Ευρώπη. Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Δεύτερον, το, η ολοκλήρωση της διαδικασίας της εύκτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την κύρωση της Συμφωνίας περί αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ε, αποχώρησης και από την ευρωπαϊκή πλευρά. Και από αυτή την άποψη κρίσιμο βήμα είναι η συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Κροατική Προεδρία Σύμφωνα με την ε, δήλωση για τις μελλοντικές σχέσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα προσπαθήσει να διευκολύνει μια ταχεία έγκριση ε, μια συνολική εντολή του Συμβουλίου για τι διαπραγματεύσει με βάση τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και παρόλο που θα μα ε, λυπήσει η αποχώρηση ενό κράτου μέλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ε, μια κοινή μακρά ιστορία. Και αυτό θα πρέπει να είναι το νέο σημείο αφετηρία για τη δημιουργία στενών σχέσεων στο μέλλον που θα εδράζονται στο στα αμοιβαία συμφέροντα, το σεβασμό και ισότιμες ηθίκε ανταγωνισμού, ιδιαίτερα στο εμπόριο, την ασφάλεια και άλλες τομέακε πολιτικές. Βέβαια, η μεταβατική περίοδο των 11 μηνών είναι εξαιρετικά βραχία και θα χρειαστεί τεράστια καλή βούληση και εργώδει προσπάθειε για να διεκπαιρεώσουμε αισίω τι διαπραγματεύσει αυτέ και να καταλήξουμε σε μια καλή εποφελή συμφωνία και για τι δύο πλευρέ. Κυρίε και κύριοι, τρίτον, η διοργάνωση της Συνόδου Κορυφής ε, στο Ζάγκρεπ, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων και η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία είναι επίσης προτεραιότητές μας. Δεν κρύβουμε την ε, φιλοδοξία μας να επιτύχουμε την υποστήριξη των κρατών μελών για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τις δύο αυτές χώρες. Η επόμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι προτάσεις της για τη βελτίωση της μεθοδολογίας των ενταξιακών διαπραγματεύσεων θα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Για την αξιοπιστία της ε, πολιτικής μας για τη διεύρυνση είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε τις αρχές του σεβασμού των, κριτικών, των ε, πολιτικών κριτηρίων, των κριτηρίων αναφοράς και των μεμονωμένων πρόοδων όλων των υποψηφίων χωρών με βάση τα αποτελέσματά τους ε, η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον απότερο στόχο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και αυτό θα πρέπει να είναι και ο κεντρικό άξονα τη πολιτική διεύρυνση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερω που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τον Οκτώβριο ψήφισμα στηρίζοντα την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, υπογραμμίζοντα τη σημασία που έχει η διεύρυνση τόσο για τι υποψήφιε χώρε όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το ψήφισμα αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, επανεπιβεβαίωσε την προσήλωσή του σε μια αξιόπιστη πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σύνοδο Κορυφή του Ζάγκρεπ με τα Δυτικά Βαλκάνια που θα γίνει το Μάιο θα λάβει χώρα 20 χρόνια μετά την πρώτη Σύνοδο Κορυφή του Ζάγκρεπ που διάνοιξε τις ε, ευρωπαϊκές προοπτικές ε, των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και επίσης άνοιξε το δρόμο για τις συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης. Μεταξύ εκείνων των χωρών βρισκόταν τότε και η Κροατία, που στο μεταξύ είναι η μόνη χώρα που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, σήμερα η Κροατία προεδρεύει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικό μας παράδειγμα λοιπόν δίνει στην ε, επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής του Ζάγκρεπ μια συμβολική συμπληρωματική αξία. Και γι' αυτό στη διάσκεψη κορυφής του Ζάγκρεπ θέλουμε να στείλουμε ένα στεναρό μήνυμα προς τους εταίρους μας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που βρίσκονται ακόμη σε ένα είδος ε, ευρωπαϊκού προθαλάμου. Και θέλουμε να τους πούμε ότι αν συνεχίσετε όλες τις μεταρρυθμίσεις και εκπληρώσετε όλα τα κριτήρια της ένταξης, η ευρωπαϊκή σας προοπτική δεν θα τεθεί ένα αμφιβόλο και θα είστε ευπρόσδεκτοι. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε τους στόχους σας χάρη στη συμμετοχή σας σε ευρωπαϊκά σχέδια, στην ε, ένταξή σας σε δίκτυα υποδομών, χάρη σε έναν τακτικό πολιτικό διάλογο στα υψηλότερα κλιμάκια και στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο και με την πραγωγή των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών. Τέταρτον, η διοργάνωση της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Και μάλιστα θα αγγίψουμε στο έργο αυτό το συντομότερο δυνατό, ώστε με βάση την πρόταση του Συμβουλίου θα συνάψουμε δύο οργανικές συμφωνίες, το συντομότερο δυνατόν, και ε, προσβλέπουμε στην εξασφάλιση της άμεσης έναρξης της διάσκεψης αυτής για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι λοιπόν σημαντικό Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν κτήμα του στόχου στόχους της διάσκεψης αυτής και να εκπροσωπούνται ισότιμα στη διάσκεψη. Η διάσκεψη αυτή θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών, των εθνικών κοινοβουλίων και μια ευρύτερη συμμετοχή και των Ευρωπαίων πολιτών και ιδιαίτερα των νέων. Θα πρέπει να είναι ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς η διάσκεψη και να ε, προσανατολιστεί σε ζητήματα που προκύπτουν από το στρατηγικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους πολιτικούς προσανατολισμούς της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως ε, να επικεντρωθεί στα θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν κυρίως τους Ευρωπαίους πολίτες. Και χαιρόμαστε που η Επίτροπος από την Κροατία, η Ντούμπραφκα Σούιτσα, είναι επιφορτισμένη ε, εκ μέρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την προετοιμασία αυτή τη διάσκεψη. Η διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη θα είναι μια νέα ευκαιρία να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στου πολίτε και να αντιληφθούμε ε, μέσω του διαλόγου τι ε, επικρίνουν οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε γιατί αυτή η αυξανόμενη διαφορία των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αίσθηση της αποξένωσης. Τι οδήγησε στο Brexit και τη, στην έξαρση του σκεπτικισμού. Θα πρέπει να δούμε γιατί ενισχύθηκε ο λαϊκισμός και αυτή η δυσαρέσκεια απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να τα αντιληφθούμε από κοινού όλα αυτά για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε και να αλλάξουμε. Επίση, θα δώσουμε την ευκαιρία με τη διάσκεψη στου πολίτε να μα πούν τι είδου Ευρώπη θέλουν, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στι προσδοκίε του. Κυρίε και κύριοι, η Κροατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου με τέσσερις ομάδες προτεραιοτήτων. Και αυτές είναι οι εξή. Η Ευρώπη που αναπτύσσεται. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε μια ισότιμη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες όλων των κρατών μελών και των περιφερειών τους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών που δημιουργούν ε, ποιοτικές ε, συνθήκες εργασιακές και βιωτικές και συμβάλλουν στην ε, προστασία του περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Μάλιστα στο Συμβούλιο θα το συζητήσουμε σε πολλές περιπτώσεις ανάλογα με την εμβέλεια και το πεδίο εφαρμογή και θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε κατάλληλη χρηματοδότηση της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας. Και Γι' αυτό θα θέλουμε να εξασφαλίσουμε και την κλιματική ουδετερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2050. Η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και η προώθηση της ψηφιοποίησης, οι επενδύσεις στην καινοτομία και την έρευνα, η ποιοτική και διαβίου κατάρτιση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα ανταποκρίνονται στις ε, ανάγκες ε, εργασιακές του μέλλοντος. Όλα αυτά είναι σημαντικά διακυβεύόμενα της ενίσχυσης της ε, ανταγωνιστικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης απαραίτητη συνιστόσα της ανάπτυξης είναι η ανταγωνιστικότητα. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να αναπτύξουμε την αγορά εργασία μας που θα προσανατολίζεται στις ανάγκες των καιρών και στην ψηφιακή ε, στην ψηφιακή επανάσταση, αλλά θα λαμβάνει υπόψη και τις δημοκρατικές αλλαγές. Γι' αυτό θέλουμε και δημογραφικά μέτρα που να δημιουργούν ε, μια πιο ζωηρή κοινωνία. Η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να αξιοποιεί το δυναμικό, το ανθρώπινο, αλλά και των υποδομών. Και η σωστή διασύνδεση είναι από τις σημαντικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής των κρατών μελών. Γι' αυτό θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω τις υποδομές μεταφορών, ενέργειας ε, και ψηφιοποίησης προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Και γι' αυτό θέλουμε να φέρουμε πιο κοντά τους πολίτες χάρη στην παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Αυτοί οι δεσμοί ε, ε, αντανακλούν την ισχύ μας και την κοινότητά μας. Κυρίες και κύριοι, ο τρίτο άξονα προτεραιοτήτων μα είναι η Ευρώπη που προστατεύει, γιατί μόνο μια ασφαλή Ευρώπη μπορεί να εξασφαλίσει ένα ειρηνικό περιβάλλον για του πολίτε τη. Και από αυτή την άποψη, η αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και μια αυξανόμενη αθεκτικότητα προ τι εξωτερικέ απειλέ και τι υβριδικέ και κυβερνόπειλε έχουν ζωτική σημασία. Η υλοποίηση μια συνολική λύση για μια βιώσιμη και αποτελεσματική πολιτική μετανάστευση και ασύλου είναι κοινό μα στόχο θα παραμείνουμε εστιασμένοι στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσής μας ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης με βάση τις κοινέ μας αξίες, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Ως εκ τούτου, η έγκριση της, των νέων στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών στον χώρο ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης θα είναι προτεραιότητά μας. Το κράτος δικαίου είναι πρωταρχική αξία και θεμελιώδης αρχή της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επιδιώξουμε λοιπόν μια συνολική προσέγγιση που θα προστατεύει και θα προωθεί το κράτο δικαίου, ενώ θα ενισχύει ταυτόχρονα το διάλογο και την ενότητα των κρατών μελών. Τέταρτη προτεραιότητα. Μία Ευρώπη με βαρύτητα που θα ασκεί επιρροή. Κανένα μεμονωμένο κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνο του τι διεθνεί απειλέ μας, λοιπόν, η ενότητά μας λοιπόν είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας. Θα πρέπει να αποφαινόμαστε με νέα φωνή πιο συχνά και πιο ηχηρά και να επιβεβαιώνουμε τον παγκόσμιο μας ρόλο σε αυτόν τον πολυπολικό κόσμο. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε έναν ανοιχτό διάλογο με τους βορειοαμερικανούς εταίρους και συμμάχους μας και η φιλοδοξία μας να γίνουμε παγκόσμιος παράγοντας θα πρέπει να συνοδευτεί από την παράλληλη παράλληλη ανάπτυξη των ικανοτήτων και των μέσων μα για κοινή δράση, ακόμη και τη άμυνά μα, παρόλα αυτά συμπληρωματικά με τον ΝΑΤΟ. Επίση, θα πρέπει να ε, διατηρήσουμε τι ευρωπαϊκέ μα σχέσει με την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία και την Ιαπωνία και άλλε μεγάλε δυνάμει, βάσει του αμοιβαίου σεβασμού, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε την πολυμέρεια και τη διεθνή τάξη βάσει κανόνων. Σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτικών από την κλιματική αλλαγή μέχρι το εμπόριο και την ε, πυρηνική ε, ανάπτυξη, ε, την ανάπτυξη των πυρηνικών, έχουμε τη μοναδική ικανότητα να καταλήξουμε συμβαστικές λύσεις και να διαθετήσουμε κρίσεις. Οι εντάσεις στην Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση ασφάλειας και πολιτικής στο Ιράν και το Ιράκ ή οι νέες προκλήσεις στον Περσικό κόλπο, όλα αυτά απαιτούν την ε, συνεχή ενεργό και δημιουργική μας ε, δέσμευση και συμμετοχή και, μια, και έναν ισχυρό ηγετικό ρόλο. Είμαι ε, μεγάλος υπέρμαχος, είμαστε μεγάλοι υπέρμαχοι του, των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και από τους μεγαλύτερους δωρητές της αναπτυξιακής βοήθειας. Και αυτό έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στις χώρες της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού. Κατά τη διάρκεια της κρατική Προεδρίας θα διοργανώσουμε και διάσκεψη κορυφή τη Ανατολική Γειτονία. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζουμε, αντιμετωπίζει πολυάριθμες προκλήσεις. Ο κόσμος μας γίνεται καθημερινά όλο και πιο περίπλοκος και οι απαιτήσει όλο και περισσότερες. Έχουμε πολλέ. Ε, πολλούς παράγοντες που προφέρουν μερικές φορές ε, εύκολες και άμεσες απαντήσεις που πολύ συχνά όμως στηρίζονται σε παραπληροφόρηση. Οι προσδοκίες των πολιτών μας αυξάνονται. Θα πρέπει να βρεθούμε κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες, να αφουγκραστούμε τι ανησυχίε του και να δώσουμε κατάλληλε απαντήσει στον προβληματισμό του. Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε κάτι περισσότερο για του Ευρωπαίου πολίτε. Και για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση, θα πρέπει να προωθήσουμε την ισότητα, την αλληλεγγύη, να αποφύγουμε του αποκλεισμού και να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία, που είναι η βασική μα αξία στο παγκόσμιο προσκήνιο. Και όπως λέει και το σύνθημά μας, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη σε ένα κόσμο με προκλήσεις. Σας ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστούμε κύριε Πλένκοβιτς. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας αυτή. Καλύψατε πάρα πολλά ζητήματα από το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δώσω τώρα το λόγο στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φοντελάιν. Ευχαριστώ για την παρουσία της εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι με μεγάλη χαρά Κύριε Πρωθυπουργέ, που σας ξαναβλέπω εδώ στις αρχές της Κροατικής Προεδρίας, πριν από λίγες μόνο μέρες το σώμα των επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματικά δέχθηκε την καταπληκτική αυτή κροατική φιλοξενία. Περάσαμε μια καταπληκτική ημέρα στην Κροατία, όπου καταφέραμε να δούμε πάρα πολλές διαφορετικές πτυχές του πολιτισμού και της παράδοσής σας, όλα αυτά τα οποία έχει συνεισφέρει η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά η τελετή στο Εθνικό Θέατρο της Κροατίας του Ζάγκρεπ ήταν καταπληκτική και πραγματικά καταδεικνύει τον ενθουσιασμό με τον οποίο εργάζεται η Κροατία στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι θα πρέπει ε, να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μπορούμε ακόμα αυτή τη στιγμή στον οίκο τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία να ακούμε πραγματικά τι προτεραιότητε Κροατική Προεδρία. Αντρέη, γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα προσφυλέ σε σένα. Και δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να πούνε ότι πραγματικά έχουν, ε, έχουν υπάρξει ασκούμενοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αργότερα γίνανε ευρωβουλευτές και έπειτα επιστρέφουν στο Στρασβούργο ως πρωθυπουργοί και μάλιστα προεδρεύοντες της, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρητήρια λοιπόν, Αντρέη. Κατά κάποιο τρόπο η στεδρομία σου αυτή καθρεφτίζει πραγματικά την, το καταπληκτικό ταξίδι το οποίο ακολούθησε η δική σου η χώρα, η Κροατία. Όπω είπε, μόνο μέσα σε τρει δεκαετίε η Κροατία κατάφερε να περάσει από συνθήκε αιματοχυσία στην Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αύριο θα έχουμε την ε, επέτειο των 28 ετών από τότε που η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναγνώρισε την εξαρτησία της Κροατίας. Ουδής όμως τότε θα μπορούσε να φανταστεί πόσο μακριά και πόσο γρήγορα θα προχωρούσε η χώρα αυτή. Και αυτό έχει να κάνει με τη βούληση του δικού σου του λαού, των θυσιών που έχουν κάνει έχει να κάνει με τη δέσμευσή του στι ευρωπαϊκέ αξίε και έχει να κάνει και με την αποφασιστικότητά του να ενταχθούν σε μια ένωση ευημερία και ειρήνη. Λοιπόν, του επόμενου λοιπόν έξι μήνε θα χρειαστούμε αυτή την ενότητα, αυτή τη συλλογικότητα, την ενέργεια και την αποφασιστικότητα για την οποία είναι διάσημοι οι Κροάτε. Θα πρέπει πραγματικά να βρούμε κοινέ λύσει για κάποια ζητήματα τα οποία μα δίχασαν στο παρελθόν, όπω για παράδειγμα η μετανάστευση. Θα πρέπει να ασχοληθούμε προφανώ με τον τομέα αυτόν, αλλά θα χρειαστούμε και τη συλλογικότητα αυτή, την ενότητα αυτή για να αντιμετωπίσουμε το Brexit, τι διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα διεθνή ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε και θα χρειαστούμε και την ενέργειά σα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει με επιτυχία όλη αυτή τη μεταβατική περίοδο όσον αφορά την οικονομία και την ενέργεια. Και χαίρομαι πάρα πολύ που οι προτεραιότητε τη Κροατική Προεδρία πραγματικά αντικατοπτρίζονται στου τέσσερι αυτού πυλώνε που έθιξε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργό. Λέγεται ότι χρειαζόμαστε μία Μα λέτε εσεί, μάλιστα, στο σλόγγαν τη Προεδρία, ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη σε ένα κόσμο προκλήσεων. Και όντω βλέπουμε ότι οι προκλήσει αυτέ εντείνονται μέρα με την ημέρα και νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή μια επικοδομητική δύναμη προκειμένου να καταφέρουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυνάμεις της ε, καταστροφής. Όσο αντιμετωπίζουμε συνθήκες ε, βίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ε, βία αυτή ουσιαστικά συνεχώς θα επαναλαμβάνεται και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βασιστούμε στην πραγματική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει μια πολύ ισχυρή δυναμική, ε, διπλωματική δύναμη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε το διάλογο, ακριβώς επειδή έχουμε πάρα πολλές θετικές σχέσεις με πάρα, πολλούς, ε, με πάρα πολλές χώρες και πάρα πολλούς παράγοντες στην Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι ακριβώς επειδή έχουμε έναν ε, ρόλο ιδιαίτερα σταθεροποιητικό, ιδίω όσον αφορά το Ιράκ και όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι παράγοντε μα δείχνουν εμπιστοσύνη. Νομίζω όμω ότι στο διεθνέ προσκήνιο θα πρέπει να καταφέρουμε να ενισχύσουμε τη θέση μα, να ενισχύσουμε τη θέση μα ω τον πιο σημαντικό εταίρο σε παγκόσμιο προσκήνιο, θα πρέπει να δεσμευτούμε περισσότερο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, να λάβουμε περισσότερε ευθύνε, θα πρέπει να ενισχύσουμε του δεσμού μα με την Αφρική και θα πρέπει να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την οικονομία και στην Αφρική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουμε μάλιστα και μία συνεδρίαση των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με παράγοντες της ε, Αφρικής στα πλαίσια της ε, Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής που θα λάβει χώρα και θα διοργανωθεί αυτό και κατά τη διάρκεια της δικής σας Προεδρίας. Οι επόμενοι έξι μήνες θα είναι πάρα πολύ σημαντικοί όμως και για τις σχέσεις που θα έχουμε με τις Βαλκανικές χώρες. Το είπες και εσύ, Αντρέη. Η Κροατία το γνωρίζει αυτό καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον πόσο σημαντική είναι η δύναμη ισχύ τη ευρωπαϊκή προοπτική. Θα πρέπει να υπάρχουν αυτέ οι προοπτικέ, να είναι πραγματικέ προοπτικέ. Και η Κροατία το γνωρίζει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, πόσο πολύ μπορεί να προωθήσει η προοπτική αυτή τα συστήματα και τι οικονομίε μια χώρα. Η Κροατία γνωρίζει τις θετικές επιπτώσεις μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων μπορούν να γίνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να διατηρήσουμε την δυναμική αυτή προχωρώντα προ τη Σύνοδο Κορυφή του Ζάγκρεπ μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των Δυτικών Βαλκανίων. Αν πραγματικά θέλουμε η Σύνοδο αυτή, αυτή να στεφθεί με επιτυχία, θα πρέπει να καταβάλουμε πάρα πολλέ προσπάθειε. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προωθήσουμε μέσα σε επόμενε εβδομάδε την πρόταση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον εξεχρονισμό τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τι ενταξιακέ διαπραγματεύσει. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να δώσουμε και μια πραγματική χειροπιαστή ευρωπαϊκή προοπτική στους ε, εταίρους μας στην ε, Αλβανία και στη Βόρεια Μακεδονία. Έχουν καταβάλει πολλές προσπάθειες, έχουν κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να τους δώσουμε μια ειλικρινή αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκή προοπτική. Πολύ σημαντική όμως θα είναι και η συμβολή της Κροατίας στις ε, διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τις επόμενες εβδομάδες το Συμβούλιο με την Προεδρία του κυρίου Μισελ θα προσπαθήσει να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και σε ένα προπολογισμό ο οποίο θα είναι ισορροπημένο, δίκαιο και χρειαζόμαστε κυρίω και ένα προπολογισμό ο οποίο να είναι σύγχρονο, μοντέρνο. Τα επόμενα 7 χρόνια θα διαφέρουν από τα προηγούμενα 7 χρόνια τα οποία μόλι τώρα διανύσαμε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό του εξυγχρονισμού, η πτυχή του εξυγχρονισμού να στεφθεί με επιτυχία. Αυτό περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτε, αυτό ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναλάβουμε δράση, να είμαστε ω Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πιο προβεβλημένοι και ορατοί. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα αξιοπρεπή προπολογισμό, ο οποίο θα πρέπει να εξυγχρονιστεί. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για όλε τι προσπάθειε που έχετε καταβάλει εσεί εδώ. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, οι έξι μήνες της κρατική προεδρίας ήταν επίσης καθοριστικοί προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε την οικολογική και ενεργειακή μετάβαση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε απλώς μόνο για έκτακτη ανάγκη. Θα πρέπει να αναλάβουμε δράση και να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Οι εργασίε ξεκινούν ήδη από σήμερα και μετά τη σημερινή μα συζήτηση οι Ευρωπαίοι Επίτροποι θα συζητήσουν ε, της, ε, το, την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι βιώσιμε επενδύσει, καθώ επίση και το μηχανισμό και το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση. Κατά αυτόν τον τρόπο, μέσω του Ταμείου αυτού, δίνουμε τη δυνατότητα στι περιφέρειες εκείνε οι οποίε θα αντιμετωπίσουν τι περισσότερε δυσκολίε κατά την οικολογική και ενεργειακή μετάβαση να βοηθηθούν στι προσπάθειέ του αυτέ. Ξέρω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Κροατία αλλά και για πολλέ άλλε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσει αυτέ. Οι αντιπρόεδροι και Τίμερμαντ θα έλθουν εδώ πάλι στην Ολομέλεια προκειμένου να σα παρουσιάσουν όλε τι λεπτομέρειε των προτάσεων αυτών. Βασίζομαι λοιπόν στην στήριξη τη Κροατική Προεδρία για να προωθήσουμε το φάκελο αυτόν και όλου του υπόλοιπου φακέλου και όλε τι υπόλοιπε προτάσει, τι οποίε θα καταθέσουμε τι επόμενε εβδομάδε και του επόμενου μήνε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θα κλείσω με τις γλώσσες, με τις, τα, τα λόγια μίας συγγραφέως από την Κροατία Μαρία Ζαγκόρσκα, η οποία είχε πει ότι εκεί που υπάρχει ενότητα υπάρχει και ελευθερία. Και αυτό πράγματι πάντοτε ίσχυε για την Ευρώπη όταν υπάρχει ενότητα και η ιδιαιτερότητα είναι ότι πρόκειται για εθελούσια ενότητα στην Ευρώπη, τότε υπάρχει και ισχύσια. Και είμαι πεπισμένη πως η Κροατική Προεδρία θα είναι μια Προεδρία της Ενότητας, θα είναι μια προεδρία της ισχύω ε, της Ευρώπης, θα είναι μια προεδρία ε, που θα προωθήσει τους θεσμούς γιατί όπως είπατε θα προωθήσετε μια πιο ισχυρή Ευρώπη σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Ας ακούσουμε τώρα τους πρόεδρους των πολιτικών ομάδων και ξεκινάμε με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ έχει το λόγο παρακαλώ. Welcome, Andrei Plenković. Καλώ ήρθε, Αντρέ Πλένκοβιτ. Καλώ ήρθε, Κροατία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε μαζί μα. Άκουσα και τα λόγια και τι εξηγήσει που έδωσε η Ursula Φόντερ Λάιεν ε, παρουσιάζοντα την ιστορία, στην ιστορία του Αντρέ Πλένκοβιτ. Και πραγματικά νομίζω ότι μα παρακινεί όλου ιδιαίτερα η ιστορία σου. Αλλά έχουμε και αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Κροατία, κάθεται δίπλα στην Ursula Φόντερ Λάιεν. Έχει μια παρόμοια ιστορία. Εξελέγει αρχικά ευρωβουλευτή και τώρα ε, έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του σώματο ε, των επιτρόπων. Και όλα αυτά έχουν ιδιαίτερο συμβολισμό για το τι σημαίνει η Κροατία ε, για μα όλου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρώπη. Αγαπητοί φίλοι, η Κροατική Προεδρία είναι μια πάρα πολύ καλή αφετηρία για αυτή τη δεκαετία. Είναι το νεότερο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση Κροατία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι ο κρατικό λαό έδειξε πως ε, ε, είναι ενδιαφέρον για, το, για την ίδια τη χώρα και χρήσιμο να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το είδαμε. Μετά το 2013 βγήκε η χώρα από βαθιά ύφεση. Ε, το 70% περίπου όλων των εξαγωγών πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 3.000 ε, περίπου κρατικέ ΜΜΕ εποφελούνται από το νέο επενδυτικό πρόγραμμα. Λίγα μόνο παραδείγματα αυτή τη πολύ επιτυχημένη κροατική ε, ιστορία. Γι' αυτό χαιρόμαστε που είναι στο πιδάλιο της Ένωσης αυτό το εξάμεινο η Κροατία η οποία δείχνει και την ομορφιά ε, της Ευρώπης. Στο Σπλίτ, ρωμαϊκή κληρονομιά, στο Ζάγκρεμπ, ρωμαϊκή αυτοκρατορία, στο Ντουμπρόβνικ, βενετσιάνικες επιρροές Νομίζω ότι αντικαθεπτρίζει λοιπόν ε, την πολυμορφία και την ομορφιά του ευρωπαϊκού πολιτισμού η Κροατία. Και το σημαντικότερο για εμά σήμερα, το είπε και η Ούρσουλα Φοντρελά, είναι ότι η Κροατία είναι ένα ανεξάρτητο κράτο. Είναι ένα ανεξάρτητο κράτο, δεν ανήκει σε καμία αυτοκρατορία, αλλά ανήκει σε μια οικογένεια. Και τη σεβόμαστε όλοι. Είναι ένα ισότιμο μέλο τη ευρωπαϊκή οικογένεια. Και νομίζω ότι αυτή η έντονη ευρωπαϊκή προοπτική αντικαθρεπτίζεται και στο πρόγραμμά σα. Ευρώπη που θα δώσει απαντήσει στι παγκόσμιε προκλήσει. Αυτό είναι το σλόγγαν, αυτό είναι το σύνθημά σα. Και πραγματικά ε, πρέπει να πούμε ότι σε αυτού του πολύ ταραχώδει καιρού που ζούμε, κανένα κράτο, αν σταθεί μόνο του, δεν έχει ελπίδε ε, και πιθανότητε να πετύχει. Έχουμε παγκόσμιε προκλήσει, έχουμε την ψηφιακή επανάσταση την ανάγκη να προσφέρουμε ασφάλεια στους πολίτες ε, και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Ε, το κλειδί είναι η ενότητα. Το είπε και η Ursula von Και θέλω να περιγράψω ε, λίγο πολύ τι εννοούμε με τη λέξη ενότητα. Για μας ενότητα σημαίνει δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, αν η Κροατία θέλει να προσχωρήσει στο χώρο του Σέγγεν, αν θέλει να είναι μέλος στην Ευρωζώνη, θα έχει την πλήρη υποστήριξή μας. Ενότητα επίση σημαίνει ευρωπαϊκή προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια. Προαναφέρθηκε και Πιστάκης Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν κοντόθωρη να μην ξεκινήσουν δηλαδή ενταξιακέ διαπραγματεύσει με Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία και εγώ πραγματικά είμαι ως ε, μέλος του ΕΛΚ υπερήφανος για το ότι υποστηρίχθηκε αυτή η πρόταση από, όλους, ε, από όλα τα μέλη του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο και θα μιλήσουμε ε, και το ίδιο θα κάνουν και οι Γάλλοι συνάδελφοί μας με τους αρμόδιους ώστε να ανοίξουν οι πόρτες, ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις. Για μας ενότητα, αγαπητοί σύντροφοι, σημαίνει όλοι για έναν και ένας για όλους ε, στο διεθνές προσκήνιο. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες ε, ήμασταν μάρτυρες των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πραγματικά ήμασταν πολύ κοντά σε μια πολεμική κλιμάκωση. Ακούστηκαν ε, πολύ ηχηρέ φωνές, αλλά εμείς έχουμε υψώσει και μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό πιο ηχηρά ακόμη και, πιο, και το ανάστημά και τη φωνή μα. Και οι πρώτες εβδομάδες αυτής της δεκαετίας νομίζω είναι και μια αφύπνιση για εμάς. Ε, πρέπει να δείξουμε ότι είναι ικανή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να προχωρήσουμε με το στρατιωτικό πυλώνα της ένωση. Ε, και θα πρέπει να ξεκινήσει και η διαδικασία λήψη αποφάσεων. Ε, θα πρέπει να αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού, να μην αποφασίζονται πλέον τα θέματα ασφάλεια και πολιτική με ομοφωνία, αλλά με ειδική πλειοψηφία. Ενότητα σημαίνει επίση και ε, για το Brexit. Δική μα λέσχη, δική μα οι κανόνε. Υπάρχουν τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα σε όλες τις χώρες μέλη της Ένωσης. Ε, σε καμία περίπτωση κανείς δεν θέλει να τιμωρήσει ε, τους Βρετανούς φίλους. Κάποιοι μπορεί να το ισχυρίζονται αυτό. Όχι όμως. Ε, αν κάποιος δεν είναι μέλος της Ένωσης, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, όμως χάνει τα πλεονεκτήματα και τα προνόμια της λέσκης στην οποία είναι μέχρι τώρα. Ε, και πρέπει να ε, πείσουμε τους πολίτες ότι είναι καλύτερο να παραμείνουν εντός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα πολλές οι προκλήσεις μπροστά μας, αλλά πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Και τέλος, για το πει. θα πρέπει να έχουμε έναν επαρκή προπολογισμό που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τα αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, για να είναι πιο ασφαλής η Ένωση. Επενδύσεις επίσης στην έρευνα και την καινοτομία. Και αυτό θα βοηθήσει όλους τους πολίτες. Μην μιλάμε λοιπόν για καθαρούς εισφέροντες ε, ή ε, καθαρούς δικαιούχους. Έχουμε νέα καθήκοντα μπροστά μας που σημαίνει ότι θέλουμε και νοπό χρήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι οι προκλήσεις για την κρατική Προεδρία. Είναι Καιρός όμως ε, να δείξουν το δρόμο ε, η ε, νεότερη, η νεότερη χώρα να δείξει η ηγετική στάση και να αποδείξει ότι η Ευρώπη έχει μέλλον. Και πρέπει να σας πω ότι μπορείτε να βασιστείτε στην βοήθεια του ΕΛΚ. Ευχαριστούμε. Εξ ονόματος των Σαλιστών τώρα η πρόεδρος Γκαρσία Πέρες έχει το λόγο. Κύριε Πλένκοβιτς, ε, με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχόμαστε η εμπειρία που είχατε ως Ευρωβουλευτής ε, να συμβάλλει στην επιτυχία της κρατικής προεδρίας. Έχουμε επίγνωση το ότι διανύουμε μια ταραχώδη περίοδο που βρήθη προκλήσεων ε, αρκούν ε, τα γεγονότα και εξελίξει ε, στη Μέση Ανατολή για να μα πείσουν. Είπατε ότι είστε υπέρ τη πολυμερού προσέγγιση και τη στενή συνεργασία με τον είπα το εκπρόσωπο. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί έτσι θα μπορέσει η Ένωση να μιλά με μια φωνή στο διεθνέ προσκήνιο. Επίση, ε, υποστηρίζουμε την προσήλωσή σα στην πολιτική διεύρυνση και την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Οι προτεραιότητες ε, του προγράμματός σας μεταξύ άλλων ήταν ε, μια Ευρώπη που προστατεύει και σε αυτό τον τίτλο θα θέλαμε ε, να αναγνωρίσετε μεταξύ άλλων τη σημασία της μετανάστευσης για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και της διατήρησης του κράτους πρόνοιας. Ναι, κύριε Πλένκοβιτ, χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που να προστατεύει. Μια Ευρώπη όμω που προστατεύει τι σημαίνει. Σημαίνει και αλληλεγγύη, σημαίνει και κράτο δικαίου, η Ευρώπη πρέπει επίσης, ε, αν θέλουμε να ε, είναι μια Ευρώπη που προστατεύει, να προστατεύει και τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, να τους ε, φιλοξενεί με πολύ καλούς όρους, να προστατεύει επίσης τους πολίτες της Ένωσης κατά του αποκλεισμού της ανεργίας ή των διακρίσεων λόγω φύλου. Θα σας ζητήσουμε λοιπόν να δείξετε μεγαλύτερη φιλοδοξία και για την οικοδόμηση της κοινωνικής Ευρώπης που ε, τόσο αναγκαία είναι. Ας είμαστε ειλικρινεί. Με τη διοργάνωση διασκέψεων απλά και μόνο δεν μπορούμε να κλείσουμε για παράδειγμα το μυστολογικό άσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Να πάψει να υπάρχει βία σε βάρος των γυναικών ή φτώχεια ε, μεταξύ παιδιών. Θέλουμε να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την καινοτομία, τη διαβίου μάθηση, ναι. Αλλά χρειαζόμαστε και ένα πραγματικό σχέδιο δράση για να υλοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικό Πυλώνας ε, και να γίνουν πράξη ε, τα κοινωνικά δικαιώματα. Λυπούμεθα που στο πρόγραμμά σας δεν αναφέρετε ε, την εγγύηση για τα παιδιά, τον κατώτατο μισθό, πραγματικά μέτρα καταπολέμησης της φτώχειας. Ελπίζουμε να συμπεριληφθούν τέτοια μέτρα και δράσεις ε, στο πρόγραμμά σας στη διάρκεια της Προεδρίας σας και για την ε, ε, νομισματική πολιτική. Η ασφάλιση, το επίδομα εργασίας δεν επαρκεί αυτό το οποίο προτείνεται γιατί θέλουμε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας σε περίοδους κρίσης με τα κατάλληλα μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν να νομοθετήσουμε εκεί που είναι δυνατόν να νομοθετήσουμε εκφράσατε την προσήλωσή σας για να πετύχετε συμφωνία ε, σε ένα νέο πολιτές νοσομικό πλαίσιο και αυτό ε, μας βρίσκει βέβαια σύμφωνους. Η πρόταση όμως πρέπει να είναι στο ύψος ε, της πρότασης που κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έχουμε πει και επαναλάβει πολλές φορές. Δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα με λιγότερα. Το έχουμε πει. Και για να πετύχουμε τους στόχους του φιλόδοξου θεματολογίου μας θα πρέπει να έχουμε ε, τρεις άξονες το ΑΕΠ υπάρχει ένα επαρκέ ποσοστό, να έχουμε ίδιου πόρου και να έχουμε και μια μεταρρύθμιση των φορολογικών κανόνων. Και γι' αυτό θα προασπίσουμε ε, ένα νέο χρυσό κανόνα στο σχέδιο, στο σύμφωνο μας σταθερότητας και ανάπτυξη, για την υποστήριξη και τόνο των βιώσιμων επενδύσεων στα κράτη-μέλη. Δεν πρέπει να απογοητεύσουμε τι προσδοκίε των Ευρωπαίων πολιτών με κενές ε, υποσχέσει σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο. Απαιτείται και κατάλληλη χρηματοδότηση δεν θα σα κρύψω την απογοήτευση τη πολιτική μα οικογένειας, διότι από το πρόγραμμά σα λείπει ένα σχέδιο βιώσιμων επενδύσεων σε ό,τι αφορά και το Ταμείο ε, Δίκαιης μετάβαση. Υπάρχει δέσμευση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμπερίληψη των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Εξάμεινου. Εσά ε, δεν ε, φαίνεται να σας φαίνεται προτεραιότητα γιατί δεν το έχετε περιλάβει στο πρόγραμμά σα. Πρέπει όμω να δείξετε την ίδια φιλοδοξία όπω αυτή που δείχνει η Κομισιόν με το πρόγραμμα εργασίας και εν ώψη των προκλήσεων. Αν έχετε όμως την σωστή βούληση θα έχετε την υποστήριξη τη δική μας ομάδας για την οικολογική, κοινωνική και οικολογική αλλαγή και μετάβαση που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο ομάδας Renew Europe ο πρόεδρο Ντάτσαν Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, κύριε Πλένκοβιτς, πρόκειται για την πρώτη Προεδρία της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που ενταχθήκατε το 2013 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πολύ σημαντική στιγμή για σας, για τη χώρα σας, για το λαό σας, αλλά και μια σημαντική πρόκληση. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι στην πρώτη αυτή Προεδρία δείξατε ιδιαίτερη ενέργεια και ενθουσιασμό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρετε και στον εσωτερικό κύκλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στον χώρο Σέγγεν δηλαδή, αλλά και στην Ευρωζώνη, να καταφέρετε να δείξετε παρόμοια δυναμική στάση και θα πρέπει όλες οι χώρες να μπορούν να ταχθούν στους δύο αυτούς χώρους, αυτή τη στιγμή πληρούν τα κριτήρια. Δεν θα πρέπει να διασφαλίσουμε μόνο το ότι θα ανανεωθούν οι κανόνες μας για το ευρώ, αλλά θα πρέπει το ευρώ να λειτουργεί υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών και το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι ελκυστική η Ευρωπαϊκή Ένωση για του Ευρωπαίου πολίτε. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ καθοριστική η διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη που θα μπορούσε να δώσει και νέε προπτικέ όσον αφορά τη διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω του επόμενου μήνε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει πραγματικά ένα θετικό μήνυμα προ τα Δυτικά Βαλκάνια και ότι η Σύνοδο Κορυφή του Ζάγκρεπ πραγματικά θα δραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο και θα στείλει ένα χειρό μήνυμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η μεταναστευτική κρίση που γνωρίσαμε το 2015-2016 είχε σημαντικές επιπτώσεις σε πάρα πολλές χώρες. Συντοπίσαμε ότι το σύστημα ασύλου που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Σήμερα η δική μου πολιτική ομάδα, το Renew Europe, θα υποβάλει ένα νέο σχέδιο με κάποιε νέε ιδέε προκειμένου να έχουμε ένα νέο αποτελεσματικό σύστημα ασύλου και μετανάστευση για την επόμενη δεκαετία. Α μην περιμένουμε να ξεσπάσει η επόμενη κρίση. Και ελπίζω Κύριε Προεδρεύονταν του Συμβουλίου, ότι και εσεί από τι δικέ μα ιδέε. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η μετανάστευση και οι δημοκρατικέ προκλήσει θα πρέπει να γνωριστούν περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει ω προ αυτέ να αναλάβουμε δράση. Χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρετε τι προκλήσει αυτέ στην παρουσίασή σα. Όσον αφορά τώρα το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε του επόμενου έξι μήνε πώ θα καταφέρουμε πραγματικά να εγκρίνουμε το πολιτέ σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο και θα έχετε πραγματικά κι εσεί ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διδραματίσει. Είναι πολύ σημαντικό να προωθήσετε περισσότερο τι απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα ισχυρό προπολογισμό αλλά και για τη χρησιμοποίηση των ιδίων πόρων. Ισχυρό προπολογισμό για να αντιμετωπίσουμε τι προ... προκλήσει που έχουμε μπροστά μα. Να ευχαριστήσω και εσά και το Σαρ Μισελ για όσα έχετε κάνει για τη Λιβύη, το Ιράκ και το Ιράν. Θα πρέπει πραγματικά να μπορούμε μέσω επαγρύπνηση να συμβάλλουμε στην ειρηνοποίηση τη περιοχή, στην ειρήνευση περιοχή. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή φωνή στο διεθνέ προσκήνιο και θα πρέπει να λαμβάνουμε τι προ... ευθύνε μα κάθε φορά που απαιτείται η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να καταφέρουμε να αναλάβουμε δράση προκειμένου να καθορίσουμε εμεί το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία κύριε Προεδρεύοντα και θα έχετε πραγματικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών ένα σημαντικό εταίρο τη δική μου πολιτική ομάδα, το Renew Europe. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Κέλλερ, εξ των Πρασίνων. Έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πάρα πολύ που αντλαμβάνει η Κροατία την πρώτη της Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Της εύχομαι κάθε επιτυχία. Η Προεδρία αυτή έρχεται μια πολύ καθοριστική στιγμή όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσουν ε, να νομοθετούν προκειμένου να αποκριθούν... σε όλε τι υποσχέσει που δώσανε κατά τη διάρκεια τη προκλογική εκστρατεία. Πάρα πολλά πράγματα πρέπει να κάνουμε. Να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια κλιματική κρίση που επηρεάζει του πάντε. Τώρα θα πρέπει να λάβουμε δράση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει, κάνει κάποια, έχει δώσει κάποιε υποσχέσει, τι οποίε τι χαιρετίζουμε. Χρειαζόμαστε όμω και τη συμβολή των κρατών μελών και δυστυχώ πολλά κράτη-μέλη ακόμα μπλοκάρουν, παρεμποδίζουν οποιαδήποτε νομοθετική πρόοδο θα μπορούσαμε να έχουμε στον κλιματικό τομέα. Χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την κλιματική δράση. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όντω θα αναλάβουν τα κράτη-μέλη τι ευθύνε του. Και γι' αυτό το λόγο ενθαρρύνουμε και εσά και την κυβέρνησή σα να εφαρμόσετε όλα τα μέτρα κλιματική και οικολογική μετάβαση που προβλέπονται για την Κροατία. Σε ένα άλλο τομέα που θα θέλαμε τα κράτη-μέλη να λάβουν περισσότερη δράση είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρατε και αυτό στην παρουσίασή σα. Θα πρέπει πάλι να ασκηθεί εδώ περισσότερη πίεση από τι κυβερνήσει προκειμένου να επανέλθουν στο σωστό δρόμο ορισμένε χώρε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίε αποτελούν πραγματικά πυλώνε. Ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ίδιο ισχύει και για το κράτος δικαίου και αυτό ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Και ανησυχώ πραγματικά κύριε Πρωθυπουργέ για τις εκθέσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την κροατική αστυνομία και τον τρόπο που έχουν αντιμετωπίσει ε, μετανάστες. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν φαινόμενα συστηματικής βίας, καταστροφή ε, των χώρων στέγασης ή πολλές φορές ακόμα και χρησιμοποίηση πυροβόλων όπλων. Είναι πολλέ οι μη κυβερνητικέ οργανώσει που έχουν αναφερθεί στα μέσα μαζική ενημέρωση, στα φαινόμενα αυτά και από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει η κατάλληλη έρευνα από την κυβέρνηση τη Κροατία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, αλλά γενικότερα σε οποιαδήποτε χώρα παγκοσμίω. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρει να διασφαλίσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Τα σύνορα της Κροατίας είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ό,τι συμβαίνει σε σύνορα αυτά αποτελεί και κοινή ευθύνη όλων μας. Η Κροατία είναι μια όμορφη χώρα και η πιο νέα χώρα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε λοιπόν μια καταπληκτική ευκαιρία για να δείξετε προς την υπόλοιπη Ευρώπη ποιο είναι το όραμά σας για το κοινό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Προεδρία όμως θα φωτίσει ακόμα περισσότερο τη δική σα τη δράση και πώ μπορούμε πραγματικά να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και όσον αφορά την κλιματική δικαιοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό εσεί να προωθήσετε το κράτο δικαίου την κλιματική δικαιοσύνη, θα έχετε δική μα την υποστήριξη, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε και οποιαδήποτε φαινόμενα παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Μπέτορ έχει το λόγο εξ ονόματος της ομάδας ID. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πλένκοβιτς, η σημερινή συζήτηση είναι η συνέχιση των πρώτων συζητήσεων που είχαμε ε, στο Ζάγκρεπ αρχές Δεκεμβρίου στη διάσκεψη των Προέδρων. Μας παρουσιάσετε τις ε, βασικές προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας. Πέραν όμως των ελπίδων που ε, γύρουν οι προτεραιότητες αυτές, οι τρεις αυτές προτεραιότητες έχουν και ένα πραγματικό κίνδυνο σε θέματα της διεύρυνσης. Ε, μήπως ε, είμαστε πολύ βιαστικοί γιατί θέλετε να ε, ξεκινήσετε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Ενώ γνωρίζουμε ότι οι χώρες αυτές παρόλο που είναι χώρες σύμμαχοι, φίλες χώρες με τις οποίες θα πρέπει να συνεργαστούμε, παρόλα αυτά είναι χώρες που μαστίζονται από την διαφθορά, από σαουδικά, ισλαμικά ή τουρκικά ισλαμικά κινήματα και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, ο πρόεδρος Μακρόν το Νοέμβριο είχε θέσει το βέτο της Γαλλίας για την ε, έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, κάτι που χαρακτήρισε ιστορικό σφάλμα ο πρόεδρο ε, Γιούνκερ. Και τελικά μα λέει ότι είναι έτοιμο να υποδεχθεί και τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και να μην ξεχνούμε τη Βοσνία και το Κωσυφοπαίδιο και ίσως ε, αν περάσουμε από 27 στις 29 μετά σε 31 χώρες, ίσως δεν μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το αντίθετο να την αποδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο. Αναφερθήκατε και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε λίγες μέρες ε, με το Brexit η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει πάνω από το 10% του πληθυσμού της. Οπότε θα πρέπει να επικεντρωθούμε πάλι στους ε, τομείς ε, που θα ενισχύουν τη συνεργασία με σεβασμό των ε, χαρακτηριστικών και των ε, αρμοδιοτήτων των κρατών εθνών και όχι να επιβάλλουμε όλο και βαρύτερες συνεισφορές στα κράτη-μέλη, κάτι που διχάζει ούτως ή άλλως στις Βρυξέλλες. Πολλοί στο Κοινοβούλιο Μίλησα για την πιθανότητα δημιουργία ίδιων πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το πρώτο βήμα μια μιας ε, ευρωπαϊκή φορολογία. Πολύ κακό μαντάτο για το φορολογούμενο που ε, θα, αυξάνε... θα βλέπει το φορολογικό του άχθο να αυξάνεται με ελάχιστο αντίκρισμα και αντίτιμο. Είπαμε ότι θέλουμε συζήτηση χωρίς ταμπού για τη λειτουργία και τον προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωση. Πολύ φοβούμαι ότι μερικοί θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη συζήτηση για να προωθήσουν την ένταξη, να αφισβητήσουν την, ε, την ε, ψηφοφορία με ομοφωνία ζητώντα την ειδική πλειοψηφία και θέλετε να πάμε ακόμη πιο μακριά, ενώ έχουμε διαπιστώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανίκανη να προστατεύσει τα σύνορά τη από τη μετανάστευση, είναι ανίκανη να προστατευτεί οικονομικά απέναντι στι ε, μεγάλε υπερδυνάμει, ε, η απούσα στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ, στο Ιράν. Και στην ουσία σήμερα περιοριζόμαστε απλώς να δίνουμε μαθήματα και κηρύγματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες και κράτους δικαίου στις χώρες μέλη. Το Brexit ε, θα είναι όντως πρόκληση και με νύχη και με δύο θα προσπίσει ο Πρωθυπουργό Τζόνσον τα βρετανικά συμφέροντα. Θα πρέπει όμως στο μέλλον η Μεγάλη Βρετανία να γίνει κερκόπορτα εισαγωγή αθέμητων, προϊόντων αθέμητου ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να τη σεβαστούμε. Είναι μεγάλο σύμμαχο και φίλη χώρα γείτονα η Μεγάλη Βρετανία, αλλά θα πρέπει να προσπίσουμε τα δικά μα συμφέροντα. Να υλοποιήσουμε επιτέλου μια ουσιαστική οικονομική προστασία. Αυτό περιμένουν οι λαοί από εμά. Σα ευχαριστώ, κυρία Τόμασιτ, για το ECR. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Κροατία Εξήμιση χρόνια μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά αναλαμβάνει την Προεδρία. Κατά την προσχώρησή μας ήταν σαφές ότι ως χώρα ε, σε πολλά σημεία ήμασταν αναπροετοίμαστοι και η πορεία μετάβασης σε αναπτυγμένη δημοκρατία που τηρεί τι δημοκρατικέ αρχέ, το κράτος δικαίου και την οικονομία της αγοράς, αυτή η πορεία δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Ε, είχαμε πολλές προκλήσεις αυτά τα 6,5 χρόνια όχι μόνο στην Κροατία αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεταναστευτική κρίση σε μεγάλο βαθμό ενίσχυσε την κοινωνική εξαίρεση, την απόρρεια τη σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση και οι διαφορέ στην ανάπτυξη μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθούν να είναι μεγάλε. Αλλάζει και η πολιτική εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το Brexit μα έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι αν συνεχίσουμε να αποστρέφουμε το βλέμμα από το πρόβλημα, το εδαφικό εύρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί εύκολα να αλλάξει. Είναι γεγονό ότι οι νεότερε και μικρότερε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μεγαλύτερε πιθανότητε να φέρουν τι προτεραιότητέ του ε, στο πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό όταν δεν έχουμε σοβαρέ προκλήσει, όταν έχουμε διευθετήσει τα βασικά μα προβλήματα, κάτι που δεν ισχύει δυστυχώ τώρα. Βέβαια, η Κροατία με την ιστορία της έχει επανειλημμένως ε, αποδείξει ότι είναι έτοιμη να υποστηρίξει την Ευρώπη σε δύσκολους καιρούς. Περιμένουμε λοιπόν από την κροατική κυβέρνηση το επόμενο εξάμεινο να μην έχει απλώς εορταστικό χαρακτήρα, αλλά να αξιοποιηθεί σωστά ώστε να μεταρρυθμιστούν κάποιοι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί, κάποιες απαρχαιωμένε ευρωπαϊκές πολιτικές και να ενισχυθεί η θέση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρόλο που στο παρελθόν πολύ συχνά άκουσε οδηγίες από τρίτους και αγνόησε το γεγονός ότι είναι πλήρες μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει αυθεντική πολιτική, θα πρέπει επιτέλους να δείξει η Κροατία ότι είναι φιλόδοξη, ότι έχει το δικό της όραμα και ότι είναι έτοιμα, έτοιμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε συγκεκριμένους τομείς και πολιτικές. Ελπίζω να αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή η, η κροατική κυβέρνηση. Κύριε Πρόεδρε, σε εσά, του υπουργού σα και σε όσου συμμετέχουν το σχέδιο της ε, Κροατικής Προεδρίας. Εύχομαι καλή επιτυχία το επόμενο εξάμενο. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Σίντερβαντ το ρευτολόγος ονόματος Ευρωπαϊκής Νοτικής Αριστεράς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν να στραφούμε στο νέο έτος ε, και στα καθήκοντα της ε, Κροατικής ε, Προεδρίας, θα ήθελα να μιλήσω εν συντομία για την αντιπαράθεση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι καλό που οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελευταία εβδομάδα εκ νέου μίλησαν για την ανάγκη να μην πάψει να ισχύει αυτή η πυρηνική συμφωνία, αλλά θυμόμαστε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Αποχώρησε πριν από 1,5 χρόνο χρόνο η ε, Αμερική από την Πυρηνική Συμφωνία και αυτό δείξε σε μια κλιμάκωση που πραγματικά μας οδήγησε στα πρόθυρα ενός ε, μεγάλου πολέμου και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει ε, τον επαπειλούμενο αυτό ε, πόλεμο ε, και πραγματικά δεν θα πρέπει να, καταπιάζονται, να παραβιάζονται και να καταπατώνται με αυτόν τον τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν οι βάσεις να μην χρησιμοποιούνται για την, από drones. Ε, θα πρέπει να πω τώρα ε, και στην Κροατική Προεδρία ε, για το 2020 μιλήσατε για την ψηφιακή επανάσταση, μιλήσατε και για την κλιματική αλλαγή. Έχουμε πράγματι να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις, μεγαλύτερες μετά την βιομηχανική επανάσταση και θα πρέπει επίσης να υπάρξει και μια οικολογική και κοινωνική δικαιοσύνη και γι' αυτό θα πρέπει να είναι επαρκής ο προϋπολογισμός. Μιλήσατε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχει ε, το πρόβλημα ε, με τα ποσοστά και τις διάφορους πολιτικούς στόχους και προτεραιότητες. Δεν μπορούμε να περικόπτουμε την πολιτική συνοχή ε, για μεγαλύτερα έξοδα για τον εξοπλισμό, την κούρσα των όπλων, για περισσότερη άμυνα. Θα πρέπει να σκεφτούμε και την κοινωνική συνοχή. Θα πρέπει να επενδύσουμε και σε αυτήν. Και κάτι τελευταίο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σέβεται το δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και εντό των ευρωπαϊκών συνόρων. Δυστυχώ βλέπουμε στα εξωτερικά σύνορα τη Ένωση και στην κροατική μεθόριο παραβιά των δικαιωμάτων. Έχετε λοιπόν και εσεί την ευθύνη ε, για το επόμενο εξάμεινο να προασπίσετε και το δικαίωμα των ανθρώπων στο άσυλο ε, και την ε, εφαρμογή τη μεταναστευτική πολιτική να προωθήσετε και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω να πετύχετε. Σα εύχομαι κάθε Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριο Σκόλατσικ, Μην γεγραμμένο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι στιγμής επέτρεπε σε μικρότερες χώρες όπως η Κροατία να επωφεληθούν ε, οικονομικά. Στη Γεωργία, για παράδειγμα, 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ και έλαβαν κάποια αποζημίωση με την ε, συμμετοχή τους ε, στα διαρθρωτικά ταμεία. Μάλιστα, είχαμε 1,7 δισεκατομμύρια τέτοιες ενισχύσεις για την Κροατία. Σήμερα, με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο τις προηγούμενες 10 ε, χρονιές είχε καταθέσει, εισφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 60 δισεκατομμύρια περισσότερα από ό,τι ελάμβανε, δημιουργείται ένα μεγάλο χρηματοδοτικό κενό. Οπότε οι πιο αδύναμες οικονομικά χώρες ε, θα πρέπει να ενισχυθούν με τη νέα κατάσταση. Θα πρέπει να βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης. Θα πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό συνεισφοράς των κοινοτικό προπολογισμό των πιο ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών μελών. Σα ευχαριστώ. Ακούσαμε τώρα του προέδρου ε, των ομάδων και μετά τον πρώτο γύρο ο Πρωθυπουργό Πλέγκοβιτ ε, θα κάνει μια σύντομη ε, ομιλία με σχολιασμό των όσων άκουσε. Σα ευχαριστώ και ευχαριστώ του αρχηγού των πολιτικών κομμάτων για τα σχόλια και τι παρατηρήσει του επί του προγράμματο τη Κροατική Προεδρία. Θα ήθελα να σταθώ και εγώ σε μερικά από τα σημεία που επισημάνατε. Φυσικά και προσβλέπω ιδιαίτερος ε, στην στενή συνεργασία με την ε, Ursula von der Leyen και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω να είναι αποτελεσματική και η πρώτη μήνυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως θα φροντίσουμε να είναι και στο Συμβούλιο. Και αυτή την άποψη, μια και αναφέρθηκε η μετανάστευση, προσβλέπουμε στη νέα πρωτοβουλία για το πακέτο του Δουβλίνου να βρεθεί μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ ευθύνη και αλληλεγγύη με αναβαθμισμένο κανονισμό του Δουβλίνου. Σε ό,τι αφορά το Σέγγεν και το ευρώ, αυτό είναι περισσότερο κροατική στόχη, δεν ήθελα να το συμπεριλάβω στη στόχου τη Προεδρία. Σίγουρα η κυβέρνησή μου έχει δύο βασικού στόχου. Να προσχωρήσουμε στο χώρο του Σέγγεν και ευχαριστώ την Επιτροπή Γιούγκερ για το πράσινο φω που μα έδωσε ό,τι αφορά του τεχνικού όρου και την παραπομπή τη πρόταση στο Συμβούλιο από την Επιτροπή της κυρίας Φοντερ Λάιν και εμείς ε, θα προωθήσουμε στο Συμβούλιο το στόχο αυτό. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο ευρώ, ολοκληρώνουμε το σχέδιο δράσης ε, για το δεύτερο μηχανισμό συναλλαγματικής ισοτιμία και θα ολοκληρώσουμε αυτή την πρωτοβουλία στα τέλη της Προεδρίας. Αυτή η απόφαση θα ληφθεί σε επίπεδο Eurogroup. Σε ό,τι αφορά την πολυμέρεια, τι ανθρωπιστικέ πτυχέ αλλά και τον ε, πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που ανέφερε η κυρία Καρσία. Αν διαβάσετε προσεκτικά το πρόγραμμα της κρατικής προεδρίας που σα το έχουμε μοιράσει, θα διαπιστώσετε ότι λέμε πολλά για την κοινωνική ένταξη, για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Αυτά αποτελούν ένα απόσπαστο τμήμα του προγράμματο κρατική προεδρία. Ό,τι αφορά τη μετανάστευση και την προστασία των συνόρων. Το 2015 και το 2016 η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση ήταν αναφυσβήτητα μετά το τείχο του, του Βερολίνου. Ήταν αναφυσβήτητα το πιο σημαντικό φαινόμενο που έλαβε χώρα και είχε πολιτικές διακλαδώσεις και συνέπειες όχι μόνο στην πολιτική συζήτηση σε επίπεδο θεσμικών οργάνων, αλλά είχε σημαντικές επιπτώσεις στις εθνικές συζητήσεις και πολιτικές σε όλα τα κράτη-μέλη. Ως εκ τούτου, η λύση του προβλήματος είναι να ενισχύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει με ε, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια, την αναπτυξιακή